μένει τρίμηνη θεώρηση θα πρέπει να διακρίνεται ε, από άλλες θεωρήσεις, να καταργήσουμε κάθε αμφισημία, κάθε παρανόηση. Ευχαριστούμε Πίτρο, ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε.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 Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τους κύριους Γκυλιόμ, Κίλερ, Κέλλερ, Βίλστρομ και Ταβάρες για την υποστήριξη τους αυτή την έκθεση, βελτιώνοντας την. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή Κομισιών και Συμβουλίου σε ό,τι αφορά την ε, ορολογία, η οποία θα ήταν πιο κατάλληλη. Είναι καλύτερο να μιλάμε για ε, νόμιμη μετανάστευση, ε, διότι σε ορισμένα κράτη-μέλη η παράτυπη είσοδος αποτελεί παράπτωμα. Σε πολλά κράτη-μέλη η παράνομη είσοδος ε, δεν αποτελεί αξιόπινη πράξη. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να ποινικοποιούμε αυτές τις ε, ε, καταστάσεις με γενικό τρόπο αυτό λόγο στην εισηγητική έκθεση ζητούμε από τα ε, όργανα, τα θεσμικά όργανα να αναθεωρήσουν την ε, ορολογία που χρησιμοποιείται έτσι ώστε να αναζητηθεί μια πιο κατάλληλη ορολογία για το φαινόμενο της μετανάστευσης. Το δίκτυο αξιωματικό συνδέσμο για τη μετανάστευση δημιουργήθηκε από τον 377 του 2004 του Συμβουλίου ο οποίος προβλέπει, ο κανονισμός προβλέπει ότι θα αντιπροσωπεύουν ε, κράτος μέλος, ε, κάποιο κράτος μέλος στο εξωτερικό με στόχο την ε, δημιουργία και τη διατήρηση επαφών με το φιλοξενό κράτος μέλων για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, την επανεισδοχή των παράνομων μεταναστών και την διαχείριση των νόμων, της νόμιμης μετανάστευσης. Ο κανονισμός δημιουργούσε την η ε, υπηρεσία Frontex για την ε, συνεργασία της ε, επιχειρησιακής δράσης των κρατών μελών στην διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη στην κατάρτιση των συνοριακών φυλάκων, την <clears throat> ανάλυση και την παρακολούθηση των θεμάτων έρευνας και ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων, να βοηθήσει τα κράτη-μέλη μέσω της ε, τεχνικής ε, συνδρομής στα εξωτερικά σύνορα και την ε, βοήθεια προκειμένου να διοργανωθούν κοινέ επιχειρήσεις επανεισδοχής. Η Frontex έχει σημαντική αποστολή λοιπόν. Μπορεί να επιτευχθεί όμως πιο αποτελεσματικά αν η Frontex επωφεληθεί των γνώσεων και των εμπειριών των δικτύων αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης πολύ περισσότερο, αλλά μου υπόψη είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει γραφεία ή εκπροσώπη, αντιπροσωπείες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η τροπή του κανονισμού 377-2004 έχει ως ε, στόχο να επωφεληθούν, επωφεληθεί η Frontex από τις γνώσεις και τις εμπειρίες αυτών των εξωματικών συνδέσμων. Αυτό δεν είχε προβληθεί από τον αρχικό κανονισμό. Η πρόταση τροπολογίας προτείνει επίσης πρόσβαση των, ε, στις ε, πληροφορίες μέσω της ε, Infonet, της Econet που είναι ένα ηλεκτρονικό δίκτυο πληροφοριών και συντονισμού των υπηρεσιών διαχείρισης μετανάστευσης των κρατών μελών. Ε, προκειμένου να δημιουργηθούν δίκτυα αξιωματικών συνδέσμων και για να διευκολυνθεί ο μηχανισμός υποβολής εκθέσεων σχετικών με τις δραστηριότητες των δικτύων αξιωματικών συνδέσμων. Η πρόταση βασίζεται στα άρθρα 63-3β και 66 ε, της ε, συνθήκης. Σταματάω εδώ και αργότερα θα σας παρουσιάσω περισσότερες σκέψεις μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.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 με τα διάφορα αρμόδια δίκτυα για να μπορέσει να εξασφαλίσουμε ότι το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα γνωρίζουν εγκαίρως τι δραστηριότητες αυτών των δικτύων. Συγχρόνως, χάρη στις τροπολογίε του Κοινοβουλίου, η προσέγγιση βάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα υπερισχύσει για θέματα τη μετανάστευση σε επιλεγμένες τρίτες χώρες και αναφέρομαι εις ε, την παράνομη μετανάτευση ενώ το άρθρο ε, ε, το άρθρο αναφέρεται σε illegal που σημαίνει παράνομη εγώ συνήθως μιλώ για irregular και ε, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Στοχόλμης τα δίκτυα αυτά θα συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των, ε, ε, θεμάτων που οδηγούν στην παράνομη μετανάστευση και ελπίζω ότι οι τροπολογίες θα υιοθετηθούν γρήγορα κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να επέβουμε όσο δυνατόν γρηγορότερα και να διεκπαιρεώσουμε αυτό αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, λέει η Πρόεδρος και τώρα περνάμε στους ομιλητέ εν ονόματι των ε, προελτικών ομάδων και πρώτος για το ΕΛΚ είναι ο κύριος Κοέλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε κυρίε και κύριοι συνάλφοι. Πάντοτε το Κοινοβούλιο μας υποστηρίζει τις ε, προτάσεις που ανταποκρίνονται στην ανάγκη καλύτερης διαχείριση των ε, μεταναστευτικών ροών, είτε πρόκειται για παράνομη παράτυπη, είτε για νόμιμη Σε αυτή τη δυναμική εντάσσεται και συγκεκριμένη πρόταση. Ε, τροποποίηση του κανονισμού 37 του 2004 με τη δημιουργία ενός δικτύου αξιωματικών ε, μετανάστευσης. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο συνεργασίας ε, το οποίο δεν είχε προβλεφθεί όταν δημιουργήθηκε ο μηχανισμός Frontex. Στην ε, συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για 130 τρίτες χώρες στις οποίες θα υπάρχουν αξιωματικοί σύνδεσμοι σε επαφή με τις τοπικές ε, αρχές προκειμένου να προληφθούν τέτοιου είδους μεταναστευτικές ροές η, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν έχει αντιπροσώπευση σε αυτές τις χώρες, είναι πολύ σημαντική συνεργασία με τους αξιωματικούς συνδέσμους και τη Frontex. Οι πληροφορίες των αξιωματικών συνδέσμων ε, θα χρησιμοποιηθούν από αυτούς για την ανάλυση κινδύνου και για την ενίσχυση του, της συνεργασίας μεταξύ των ε, κρατών μελών και των τρίτων χωρών η ICON.net ε, που είναι ένα ασφαλές ε, δίκτυο για τον συντονισμό των κρατών ε, μελών σε θέματα διαχείρισης μεταναστευσής επιτρέπει την χρήση κονδυλίων στο πλαίσιο του Ταμείου για τα Εξωτερικά Σύνορα. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι ο εισηγητής έκανε μια εξαιρετική δουλειά όχι μόνο επειδή έθεσε σωστά το ζήτημα, αλλά και γιατί έκανε πραγματικές ε, προσπάθειες να επιτευχθεί συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες ο κύριος Μωράζ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εποφελούμε τις ε, ευκαιρίες ε, για να μιλήσω εν ονόματι του σιώδης εισηγητών της ε, πολιτικής ομάδας των συντονιστών και θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή ο οποίος προχώρησε γρήγορα και στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και όσον αφορά για για τις τεχνικές ε, τροπολογίες ε, για να καθορίσουν πιο ακριβώς τα καθήκοντα του δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης. Βλέπουμε ότι οι δραστηριότητες αυτές ε, θα επιτρέψουν μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφενός αλλά και των διαφόρων αρμοδίων υπηρεσιών από την άλλη. Πρέπει να περιλάβουμε μία προσέγγιση που να άπτεται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως είπε η Επίτροπος και ελπίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να επιλύσουμε τις, και να καθησυχάσουμε τις ανησυχίες χωρών όπως της δικιάς μου οι οποίοι θέλουν να επιτρέψουν οι ζητούντες άσυλο να μπορέσουν να προστατευθούν. Υπάρχει ένα υπόμνημα το οποίο να αποτελεί ένα ικανοποιητικό συμβιβασμό σε μία ατέρμονα συζήτηση και ελπίζω θα υπερψηφιστεί αυτή η έκθεση. Ευχαριστώ. Τώρα για τους φιλελεύθερους, ο κύριος Σιλτσέου για δύο λεπτά. Θα ήθελα να συμφωνήσω με όλους όσους συμφωνούν με τον κύριο Ντίας Δεμέρα. Νομίζω ότι έκανε μια εξαιρετική δουλειά, κάτι το οποίο μας επέτρεψε να μπορέσουμε να συζητήσουμε ένα ιδιαίτερα περίπλοκο ζήτημα και να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς που μας ικανοποιούν απολύτως. Ως εκπρόσωπος της ομάδας των Ελευθέρων Δημοκρατών θα ήθελα να πω πως το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό διότι συμπεριλαμβάνει τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά ζητήματα μετανάστευση και μεταναστευτικών ροών. Τονίζοντα λοιπόν τα ανθρώπινα δικαιώματα, μπορούμε να εγγυηθούμε μια ουμανιστική προσέγγιση, μια ορθή προσέγγιση τόσο από πλευρά υπαλλήλων που ασχολούνται με τη μετανάστευση, όσο και από πλευρά Frontex. Εξάλλου, αυτό θα επιτρέψει να βελτιώσουμε τη συνεργασία ανάμεσα στου αξιωματικού συνδέσμου των κρατών μελών και των υπαλλήλων της Frontex. Κάτι το οποίο θα τους επιτρέψει να αποτρέψουν, να, να ε, γνωρίσουν ένα καλύτερο τρόπο συνεργασίας ε, για την διαχείριση των μεταναστευτικών δρόμων. Ε, Παρακαλώ να τελειώνετε. Η αποτελεσματική διαχείριση είναι ένα θέμα σημαντικό διότι η και θεωρούμε ότι συνεχώς και αυξάνεται και θα ανασκοπευτούν στο μέλλον. Είχατε δύο λεπτά, με συγχωρείτε, σας ε, σταμάτησα πιο πριν και θα μπορούσατε να είχατε πει και περισσότερα, με συγχωρείτε πάρα πολύ και σας ευχαριστώ. Τώρα για ένα λεπτό η κυρία Κέλλερ για την ομάδα των Πρασίνων. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή ε, Δίας Ντεμέρα για την εξαιρετική εργασία διότι πιστεύω ότι η αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης πάντοτε ήταν χρήσιμη για τις ε, απελάσεις αλλά τώρα θα επιτρέψουν να διευκολύνουμε και τους τα άτομα που ζητούν άσυλο και θα καλύψουν και μία πτυχή η οποία δεν περιλαμβάνει το καθόλου στην αρχική πρόταση. Χαίρομαι διότι μπορέσατε να δώσετε μεγαλύτερη σημασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδίω τώρα μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας όπου έχει αναβαθμιστεί η σημασία του ακόμη και αν δεν το καταλαβαίνουν όλοι. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για την εξαιρετική εργασία και ελπίζουμε ότι θα υπερψηφιστεί η πρόταση την οποία διαπραγματευθήκατε. Ευχαριστώ. Και τώρα για την Ηνωμένη Αριστερά, ο κύριος Σταβάρες για 1,5 λεπτό. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω, να συγχαρώ τον κύριο Ντεμέρα για την εξαιρετική δουλειά του. Συνεργασία και διάλογος ενέπνευσαν όλη αυτή την εργασία, χαρακτήρισαν όλη αυτή τη διαδικασία. Ιδιαίτερα στο θέμα, το ακαθόδες ε, θέμα του ε, Τη ε, ε αν πρόκειται για παράνομους ή για παράτυπους μετανάστες. Ο κύριος Ντεμέρα ήταν πάρα πολύ επικοδομητικό, πολύ δυναμικός ε, και ε, βοήθησε έτσι ώστε η ορολογία που θα χρησιμοποιηθεί να είναι πραγματικά η πιο κατάλληλη. Πολύ συχνά μιλάμε για τη μετανάστευση και συζητούμε για το κατά πόσον η, πολιτική μας θα πρέπει να είναι κατασταλτική. Η κατασταλτική πολιτική υπάρχει, βασίζεται στο Σέγγεν, στη Frontex, ε, στο ρόλο των αξιωματικών ε, συνδέσμων μετανάστευσης που τροποποιείται τώρα ε, και η κατασταλτική αυτή πολιτική ε, χρησιμεύει στον έλεγχο των συνόρων. Όμως ε, η πολιτική, η κατασταλτική πολιτική δεν αποτελεί πολιτική μετανάστευση. Αυτό το λέμε πολύ καιρό, εδώ και πολύ καιρό η αριστερά και τώρα τελευταία και η δεξιά. Οπότε, αν ψηφίζαμε την έκθεση μόνο με τέτοιου είδου ε, κατασταλτικέ ε, ιδέε δεν θα ήταν δυνατό. Αλλά ε, η, καταλήξαμε ε, σε μια συμφωνία με το Συμβούλιο. Δεν πάει τόσο μακριά όσο θα θέλαμε, αλλά είναι μια συμφωνία. Ευχαριστώ ε, ε, για την, ομάδα της Ελευθερίας και Δημοκρατίας, ο κύριος Νούταλ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ένα από τα θέματα που θέλουμε να ελέγξουμε είναι ποιος μπορεί να εισέρχεται και ποιος όχι σε μία χώρα. Αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αναθέσει το καθήκον αυτό σε πρόσωπους γραφειοκράτες στις Βρυξέλλες και αυτή τη στιγμή υπάρχουν ε, φτωχά άτομα τα οποία ε, αποθούνται και δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να ρυθμίσουμε. Επίσης έχουμε ένα σύστημα δύο ε, κατηγοριών εις την ε, Αγγλία. Αν προέρχεστε από την Αυστραλία ή ε, οπουδήποτε ορισμένες χώρες έχετε ένα ανώτατο όριο εισδοχής ενώ από άλλες χώρες μπορεί να έρθει οποιοδήποτε. Παραδείγματο χάρη η Ρουμανία μπορεί να δίνει εκατοντάδες χιλιάδες ε, εθνικότητα σε ε, άτομα που εισέρχονται στη χώρα της το οποίο είναι μια γελιότης ε, δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να αναθέτουμε στους γραφειοκράτες παλίλους αυτή την εργασία γιατί κάθε χώρα θα έπρεπε να μπορεί να ελέγξει ποιος εισέρχεται ή όχι στη χώρα του και θα ήθελα να απορρίψει αυτή την έκθεση Ευχαριστώ. Υπάρχει μία ερώτηση της κυρίας ε, Μόρβαη. Ε, θέλετε να την ακούσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον ε, συνάδελφο ο οποίος αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Άγγλοι εργαζόμενοι λόγω της μετανάστευσης. Πρόκειται από μια χώρα, την Ουγγαρία, όπου, από όπου δυστυχώς πολλοί οδηγούνται στην, στο να μεταναστεύσουν στην Αγγλία είτε ως ε, νοσηλευτές είτε ως ιατροί ή ακόμα και εξειδικευμένοι εργάτες ε, Φυσικά το, και αυτό συμβαίνει λόγω του ότι το επίπεδο των μισθών στην Ουγγαρία είναι πολύ χαμηλό για τους ε, εργαζόμενους αυτούς. Κλείνει το μικρόφωνο της ομιλήτριας. Εάν θέλουν αυτοί οι εργαζόμενοι να έρθουν στην Αγγλία και έχουν ανάγκη τις ειδικότητές τους, είναι ευπρόσδεκτοι. Αλλά τι γίνεται στην περίπτωση όπου είναι κορεσμένη η αγορά και δεν μπορούμε να δεχτούμε πλέον αυτούς τους εργαζόμενους. Νομίζω ότι αυτή η τακτική είναι σφαλμένη και θα δώσω ένα παράδειγμα. Ε, ένας ε, οδηγός ταξί που με πήγε στο αεροδρόμιο σήμερα μου είπε ότι κορεύει να χάσει τη δουλειά του λόγω ότι έχουν φτάσει Πολωνοί που εργάζονται ως οδηγοί ταξί. Αυτό δεν είναι σωστό. Ευχαριστώ. Τώρα προχωράμε στο κατάλογο μιλητών και θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον κύριο Κλέης για 1,5 ε, λεπτό σαν ανεξάρτητο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όταν θέλουμε να καταπολεμήσουμε την παράνομη μετανάστευση θα ήθελα να πω ότι εγώ είμαι υπέρ εάν αυτοί οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μπορούν να καταστήσουν πιο αποτελεσματική την Frontex με βρίσκει σύμφωνο. Αλλά θέλω να τονίσω πως ε, δεν θα πρέπει να χανόμαστε μέσα σε δεδάλους γραφειοκρατικούς και να μην χάνουμε το, να βλέπουμε το δέντρο και να χάνουμε το δάσος. Το ζήτημα της μετανάστευσης είναι ένα πολιτικό ζήτημα το οποίο απαιτεί πολιτική βούληση προκειμένου να εξευρεθούν λύσεις. Σήμερα διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν χώρες όπως το Βέλγιο, ε, παραδείγματο χάρη, το οποίο ανταμείβει τους ε, παράνομους ε, μετανάστες ε, χορηγώντας τους άδεια παραμονής. Δεν καταπολεμάμε με αυτόν τον τρόπο την λαθρομετανάστευση, του αντίον την ενθαρρύνουμε. Και μπορούμε να έχουμε περισσότερους αν θέλετε αξιωματικούς συνδέσμους και περισσότερους υπαλλήλου στην Frontex εάν δεν υπάρχει πολιτική βούληση προκειμένου να επιληθεί το ζήτημα και δεν θα μπορέσουν αυτοί οι υπάλληλοι να επιλύσουν το πρόβλημα και επίσης να μην μιλάμε για παράνομη μετανάστευση αλλά για παράτυπη. Ε, δεν καταλαβαίνω πολύ καλά όμως ε, πώς ε, επιθυμούμε με τον τρόπο αυτό να μπορέσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα βαφτίζοντάς το με ένα άλλο όνομα. Πρέπει να λέμε λοιπόν τα σίγα σίκα και τις κάποιες κάθε πρόκειται για παράνομη μετανάστευση. Τώρα έχουμε τους επόμενους ομιλητές που έχουν εγγραφεί και πρώτος ο κυριος Παπαδικολάου για δύο μισή λεπτά. διαχειριστούμε τις μεταναστευτικές ροές νόμιμες και μη νόμιμες και παράνομες. στην προσπάθεια που κάνουμε να συντονιστούμε και να δείξουμε εμπράκτως την αλληλεγγύη μας μεταξύ των κρατών μελών χρησιμοποιούμε ακόμη καλύτερα όλα τα εργαλεία που διαθέτουμε. δημιουργήσαμε το δίκτυο αξιωματικών συνδέσμων για τη μετανάστευση ε, υπόθηκε και προηγουμένως περίπου 130 χώρες ε, αφορά το δίκτυο αυτό και μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε καλή πληροφόρηση. Δημιουργήσαμε τη Frontex, δημιουργήσαμε πρόσφατα την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για το Άσυλο, ε, προχωράμε συμφωνίες για την επανεισδοχή, αξιοποιούμε όλα τα ευρωπαϊκά ταμεία που διαθέτουμε και τα ενισχύουμε όσο μπορούμε χρόνο με το χρόνο. Το γεγονός ότι πλέον φτάνουμε στο σημείο να αξιοποιούμε αυτά τα εργαλεία και να τα να τα συνδυάζουμε, να βλέπουμε δηλαδή ποιες είναι οι ανάγκες Frontex, να συνδυάζουμε με το δίκτυο ε, των αξιωματικών συνδέσμων. να συνδυάζουμε κάθε μέσο και κάθε εργαλείο που διαθέτουμε ακόμη πιο στενά αυτό και μόνο δείχνει ότι προχωράμε ακόμη πιο αποτελεσματικά. βεβαίω δεν λέει κανεί ότι ε, έχουμε φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο όταν κανείς βλέπει ότι στην ελλάδα έχουμε 90% παράνομη είσοδο των λαθρομεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό και μόνο δείχνει ότι έχουμε πολλά να κάνουμε. αυτή η συνεργασία όμως και οι δυνατότητες που έχουμε αναδεικνύει ότι μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο Μα δίνει τη δυνατότητα να είμαστε αισιόδοξοι στο βαθμό που μπορούμε στο ότι η ευρώπη έχει τις δυνατότητες και με την αλληλεγγύη και τη στενή συνεργασία όλων μας θα μπορέσουμε να έχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στη συνέχεια. κυρία επίτροπε μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα στηρίζουμε κάθε τέτοια προσπάθεια της επιτροπής μην έχετε καμία αμφιβολία ότι σε κάθε τέτοια πρωτοβουλία σας θα είμαστε αρρωγοί. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο επόμενος είναι ο κύριος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε η ε, οι υπάλληλοι της Frontex και ε, των παραμεθορίων φυλακίων κάνουν μια πολύ σοβαρή εργασία για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης η οποία εξ αρχής πρέπει να καταπολεμηθεί. Υπάρχουν ε, θέματα μετανάστευσης και άρα είναι καλό να λαμβάνονται μέτρα επί του συνόλου των θέμων αυτών για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε ε, τα θέματα αυτά προς όφελος όλων των λαών της Ευρώπης. Βεβαίως οι σύνδεσμοι αυτοί πρέπει να προωθηθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να μπορέσουν να συνδράμουν τη Frontex και νομίζω ότι χρειάζεται ούτως ή άλλως μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων διότι όλα αυτά θα πρέπει να συντονιστούν και να προωθηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα με τα κράτη-μέλη κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα. Ευχαριστώ και τώρα έρχονται οι ομιλητές στη διαδικασία Catch the Eye με πρώτον τον κύριο Μπουσουτήλ. Ε, ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ως ε, εισηγητής για το ζήτημα της παρόμοιας μετανάστευσης θα ήθελα να πω ότι με ικανοποιεί ιδιαίτερα η εξέλιξη του ζητήματος και η ανάπτυξη από τον εισηγητή διότι μας βοηθάει στο να ενισχύσουμε περαιτέρω την ε, Frontex. Η έκθεσή μου σχετικά με την Frontex την οποία παρουσίασα αυτόν τον μήνα αναφέρει και αυτή παρόμοια θέματα και νομίζω πως η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα μπορέσει ναι, στην επόμενη συνεδριασή της να ε, εγκρίνει την έκθεση με τις τροπολογίες. Ελπίζω λοιπόν πως ε, θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την διαδικασία και να τη φέρουμε το συντομό δυνατόν σε αίσιο πέρα. Επίσης, η ύπαρξη αυτών των αξιωματικών συνδέσμων θα μας βοηθήσουν ιδιαίτερα στο έργο μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρώση, ευχαριστώ Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή θα μπορούσε να τύχει αποδοχής, αλλά δυστυχώς τροποποιήθηκε από τροπολογίες που κατά την άποψή μας είναι περιττές, που αντικατέστησαν την ε, όρο παράνομο μετανάστη, παράνομο μετανάστη, μετανάστη από παράτυπο μετανάστη. Αυτό είναι ένα στοιχείο Το θετικό είναι ότι δημιουργείται ένα σχέδιο αξιωματικών συνδέσμων που θα λειτουργούν και σε συνεργασία με διεθνείς οργανώσεις για να προλαμβάνουν την ε, παράνομη μετανάστευση και να ε, βοηθήσουν στην επαναπρόθεση των παρανόμων μεταναστών. Η συνεργασία λοιπόν με τους διεθνείς οργανισμούς θα μπορούσε να είναι εύκολη για να αντιμετωπίσουν επίσης και τις ε, εγκληματικές οργανώσεις, την ε, αποφυγή και την ε, κατάργηση της παράνομης διακίνησης ανθρώπων είναι κάτι που πρέπει να πετύχουμε ούτως ή άλλως. Και τώρα ο κύριος Όμπερμαϊερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τα κράτη-μέλη έχουν καθορίσει ε, του συνδέσμους αξιωματικού για να μπορέσουν να καταπολεμήσουν την παράνομη ε, μετανάστευση. Θεωρώ ότι η συνεργασία αυτή είναι πολύ σημαντική. Χρειάζεται ανταλλαγή πληροφοριών, βελτίστων πρακτικών κατά τρόπον ώστε με τις συνεργίες αυτές να υπάρξει καλύτερος έλεγχος των συνόρων διότι η ε, Frontex δεν έχει προσωπικό για αυτό το έργο. Οπότε ε, ιδίως ε, περίπτωση ε, πτώσεων, στην περίπτωση υπηκών οι οποίοι πρέπει να επιστραφούν στην Αφρικανική Ήπειρο ή κάτι παρεμφερές υπάρχει χάος και δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε την Frontex και θα πρέπει ε, να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επέμβει καλύτερα. Ευχαριστώ ο κύριος τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η πρόταση είναι πολύ σαφής για, μα... είναι μας ότι ε, δεν είναι δυνατόν με αυτόν τον ε, τρόπο να οξύνουμε τα προβλήματα με αυτή την πρόταση. Οι εξωματικοί σύνδεσμοι θα έπρεπε να προωθούν και τα δικαιώματα των ε, μεταναστών. Επίσης είναι απαράδεκτο η λέξη παράνομη να αντικατασταθεί από το παράτυπη, διότι με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να νομιμοποιούμε κάτι το οποίο, ε, κάτι παραβαίνει το, τους νόμους. Ε, οι ευρωβουλευτές θα πρέπει να ακούσουν τη φωνή του λαού της κοινή νόμης που ε, διαφωνεί. Είναι μια καρικατούρα αυτή η έκθεση, μια καρικατούρα του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ οι στον Ευχαριστώ. Οι στον κανονισμό προωθούν και την ε, νόμιμη αλλά και την παράνομη μετανάστευση διότι υπάρχει λανθασμένη εντύπωση ότι υπάρχει ένα προϊόν ε, το οποίο ε, όταν εκτίθεται ει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό μετατρέπεται από μη ευρωπαϊκό προϊόν σε ευρωπαϊκό και αυτό ότι μπορεί να εφαρμοστεί και στους ανθρώπους. Με αυτόν τον τρόπο όμως φέρνουμε τον τρίτο κόσμο στην Ευρώπη όχι προσωρινά αλλά για πάντοτε και το έχουμε πράξει εδώ και 60 χρόνια. Ευχαριστώ. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Μορβάη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Νομίζω πως ε, θα ήταν πρέπει να βρούμε τα κατάλληλες λύσεις. Ως εκ τούτου προτείνω καθένας ε, να δικαιούται στην χώρα του να μπορεί να βρίσκει τις ε, καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας και να μην ε, συνεχιστεί αυτή η κατάσταση διότι οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι καταντούν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Οι Ούγγροι εξειδικευμένοι στον ε, νοσηλευτικό τομέα, ιατροί, μέες κλπ. είναι αναγκασμένοι να μεταναστεύσουν και μεταναστεύουν σε άλλες χώρες εντός της κοινότητας και εγκαταλείπουν την Ουγγαρία. Και η Ουγγαρία ε, παρουσιάζει ιδιαίτερη έλλειψη. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάτι προκειμένου το θέμα αυτό να μπορέσει να βρει μια λύση και να μπορέσουμε να ε, δώσουμε τις απαραίτητες συνθήκες, ε, τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας στους εργαζόμενους στις χώρες προέλευσης. Ε, και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κυρία Μάλστρομ έχει το λόγο. Αν και δεν προέκυψε από την συζήτηση άμεσα, ε, βλέπω ότι έχετε σημαντική υποστήριξη από πάρα πολλές πολιτικές ομάδες κύριε Ντεμέρα. Θα ήθελα να ε, επαναλάβω ότι χαίρομαι που τονίσατε τις διατάξεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, με αυτόν τον ε, τρόπο διασφαλίζουμε ότι όλες οι σχετικές πτυχές, ημερολαμβάνουν και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τίθενται υπό εξέταση όταν συζητούμε θέματα παράτυπης μετανάστευσης στις χώρες προέλευσης. Γιατί είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση των... Ε, μάλλον ε, έχει σχέση ή ο αριθμός των μεταναστών με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες προέλευσης. Ε, και εμείς θα συλλέξουμε τέτοιου είδους πληροφορίες για τις χώρες προέλευσης και τις χώρες με τράνζιτ. Επίση, οι εξωματικοί συνδέσμοι θα πρέπει να είναι σε συνεχείς επαφέ με τις ε, αρμόδιε αρχές των χωρών προέλευση για να καταπολεμηθεί και να προληφθεί η παράτη μετανάστευση. <clears throat> Βέβαια, είναι προφανές ότι δεν αποτελεί κανονική του αρμοδιότητα παρακολούθηση κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά σίγουρα είναι βελτιωμένο το κείμενο και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ και εσάς και τους κοιόδης ηγητές. Ευχαριστώ. Dank. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε και τώρα ερχόμαστε στον εισηγητή κύριε Ντίας Ντεμέρε. Έχετε χρόνο δύο λεπτά να δευτερολογήσετε. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για τα καλά λόγια αλλά και για την δέσμευσή σας. Παναλαμβάνω για μία ακόμα φορά την, ε, τη, τη δέσμευσή σας για την εφαρμογή αυτής της ε, έκθεσης. Ε, άκουσαν, ακούστηκαν πολλές ε, θέσεις και απόψεις. Οι περισσότερες εξ αυτών εκφράστηκαν υπέρ του έκθεσή μου. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου και τη συγκινησή μου, διότι οι παρεμβάσεις ε, πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρουσες, όπως ήταν πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις που είχαμε στην Επιτροπή και έχω συμπεριλάβει πολλά σε αυτές τις παρατηρήσεις. Θα ήθελα να αναφερθώ τώρα στην Γραφείο στήριξη ε, του Ασύλου αλλά και, τον, ε, και την, ε, τον, τον ΟΗΕ, την ύπατη αρμοστία για τους πρόσφυγες. Θα ήθελα να πω ότι το θέμα έχει τεράστια σημασία και όλοι καταβάλαμε προσπάθειες προκειμένου να πετύχουμε μια ευρύτερη συνένεση. Αγαπητοί συνάδελφοι, από μια με άποψη της κεντροδεξιάς και της ε, χριστιανοδημοκρατίας θα ήθελα να πω ότι εγώ εκφράζομαι υπέρ της έκφρασης ε, παράτυπης ε, και θα ήθελα να πω πως από νομικής σκοπιά, από σημειολογικής σκοπιά και από ισικής σκοπιά απορρίπτω τον όρο παράνομη. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους για την υποστήριξή τους και ευχαριστώ όλους όσοι έλαβαν το λόγο μολονότι ε, πολλοί εκφράστηκαν και με, ε, ε, αντίθετη άποψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έτσι ολοκληρώθηκε η συζήτηση και αύριο θα γίνει ψηφοφορία. Αγαπητοί συνάδελφοι, το επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως είναι τώρα η έκθεση της κυρίας